Okay, colleagues, thank you. Please take your seats. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ καθίστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, σας καλωσορίζω σε αυτήν την καταστατική συνεδρίαση σύσταση σε σώμα της Επιτροπής μας, όπου θα εκλέξουμε τα μέλη του Προεδρείου μας. Εγώ ονομάζομαι Κλόντ Μωράης και είμαι ο μέχρι τώρα Πρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, ΛΥΒΕ και με τα χαράς ε, προεδρεύω αυτής της συνεδρίασης. Κυρίσω λοιπόν την έναρξή της. Για τα νέα μέλη, τα οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας, να πω πως είναι μια εξαιρετική Επιτροπή. Κάνω ένα είδος ομιλίας αυτή τη στιγμή, περιμένοντας όλους σας να καθίσετε στις θέσεις σας, έτσι. Είναι τεχνικές γνωστές ε, τις οποίες ε, εφαρμόζω και θα σας λείψουν. Θα δείτε δηλαδή σε, μερικές, ε, σε λίγες εβδομάδες, όταν θα περάσουν λίγες εβδομάδες εδώ γιατί τα κάνω όλα αυτά. Ε, τώρα πια δείχνω πάντως όλοι μου λένε πιο χαλαρός, με πολύ καλύτερα. Ε, και αυτό και σχετίζεται και με τα όσα συμβαίνουν εδώ σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, Απευθυνόμενο στα νέα μέλη έλεγα ότι πραγματικά κάνατε μια καλή επιλογή, πρόκειται για μια εξαιρετική επιτροπή ε, και ήταν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή που είχε τους περισσότερους φακέλους ε, κατά την, τελευταία περίοδο αυτής της ε, θητείας και πρόκειται για μια επιτροπή η οποία πραγματικά ασχολείται με τα σημαντικότερα από τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει ήδη θα το συνειδητοποιήσετε σύντομα συμμετέχοντας στις εργασίες της. Και θα ήθελα εδώ σε ό,τι αφορά τα όλα τα μέλη, εντάξει ίσως αν όχι όλα, τα περισσότερα από τα παλαιότερα μέλη, να τα ευχαριστήσω όλα, σχεδόν όλα, γιατί ίσως κάποια να μην τους άρεσαν πολύ. Γιατί βέβαια το να αρέσουμε είναι αμφίδρομο, έτσι, δηλαδή θα πρέπει να συμφωνούν και οι δύο, ο ένας να αρέσει στον άλλο δηλαδή. Άρα λοιπόν θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους προηγούμενους συναδέλφου που συμμετείχαν σε αυτήν την επιτροπή, τα μέλη της, με τους οποίους συνεργάστηκα κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Πραγματικά αποτέλεσε ένα προνόμιο για τη δική μου ζωή το να προεδρεύσω εδώ. Ίσως να θεωρείτε ότι υπερβάλλω, αλλά όταν θα έχετε ολοκληρώσει την πενταετή σα θητεία σε αυτή την επιτροπή, πραγματικά και εσεί θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ε, πρόκειται για μια εξαιρετική εμπειρία. Ευχαριστώ ε, ε επίση εδώ το προσωπικό και ειδικότερα ε, την εξαιρετική γραμματεία που έχουμε εδώ και μας υποστηρίζει. Δηλαδή εργάζεται με πραγματικά πολύ εντατικούς ρυθμούς και νομίζω πως τα μέλη εδώ που συμμετείχαν ε, μέχρι τώρα στην Επιτροπή μας το γνωρίζω πολύ καλά αυτό. Και ε, μα ζητήθηκε δηλαδή, πλησιάζοντα ε, προ το τέλο τη θητεία, να κάνουμε κάποια πράγματα και να ασχοληθούμε με νομοθεσία σε βαθμό που καμία άλλη επιτροπή δεν είχε κληθεί να κάνει. Οπότε γνωρίζετε βέβαια πω πρόκειται για πολιτικά φορτισμένα ζητήματα. Οπότε σας ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχατε στις κοινέ προσπάθειες ε, και βέβαια βλέπω πολλά από, τους, ε, από τα παλιά πρόσωπα εδώ αλλά και πολλά νέα πρόσωπα στα οποία έχουμε καλή τύχη και ε, ειλικρινά σας λέω όσοι με γνωρίζουν ξέρω ότι είμαι ειλικρινής ε, ότι βλέπω ότι από τα παλαιότερα και από τα νέα μέλη ότι πραγματικά έχουμε εδώ πολύ μεγάλη εμπειρία που συγκεντρώνουμε εδώ μεταξύ των ε, μελών που απαρτίζουν αυτή την Επιτροπή. Πραγματικά θεωρώ λοιπόν πως θα είναι πολύ πλούσια αυτή η νέα θητεία που ξεκινάμε. Άρα λοιπόν ε, μετά από αυτήν την σύντομη εισαγωγή βλέπω πως έχετε ησυχάσει όλοι και με ακούτε οπότε σας ευχαριστώ και μπορούμε να ε, ξεκινήσουμε με τις εργασίες μας για σήμερα. Στην συνεδρίαση λοιπόν αυτή σας υπενθυμίζουμε ότι θα συσταθεί το Προεδρείο της Επιτροπής, ε, κλέγοντας δηλαδή τον Πρόεδρο και τους τέσσερις αντιπροέδρους, σύμφωνα με τον κανόνα 213, δηλαδή καταρχήν θα εκλέξουμε τον Πρόεδρο και στη συνέχεια τους αντιπροέδρους. Ε, θα ήθελα όλοι να επαληθεύσετε ότι έχετε φέρει μαζί σας τις ε, κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. αν δεν το έχετε κάνει, σας παρακαλώ να το ομολογήσετε τώρα, έτσι. Δηλαδή, να είστε ειλικρινεί, να μα πείτε αν δεν έχετε φέρει την κάρτα για να βρούμε μια λύση τώρα. Έχετε όλοι τι κάρτε σα. Έχετε βάλει με τον σωστό τρόπο την κάρτα μέσα στο μηχάνημα. Ναι, να σας πω ότι η κάρτα μου έρχεται τώρα, σε δύο ε, λεπτά θα είναι εδώ. Απάντηση του Προέδρου. Ε, εντάξει, την έχουμε ακούσει αυτή τη δικαιολογία επανειλημμένα, έχουμε ακούσει κάθε είδους δικαιολογία. Αν μα σε δύο λεπτά θα είναι εδώ, σε τέσσερα λεπτά μάλλον θα είναι. Εντάξει, πάντως θα πρέπει όλοι να φροντίσετε να έχετε τις κάρτες σας. Μετά, με βάση τον κανόνα 209 παράγραφος 7 του καταστατικού μας, θα πρέπει να ανακοινώσω ποια είναι τα απληρωματικά μέλη τα οποία θα έχουν το δικαίωμα ψήφου, δηλαδή που αντικαθιστούν ε, τακτικά μέλη. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, οπότε σας αναφέρω τα εξή ονόματα. Ρόμπερτ που ε, αντικαθιστά την ε, Άννα για το ΕΛΚ Λόραντ Βιντσέντσι που αντικαθιστά το Ραλίς ε, Μπόγκταν, Βιάτα Κέμπα για την Μάγκη Τζάκινγκ, Ρόμπερ Προύς που αντικαθιστά την Βιλάβα Βοξάντη, Αλεξάνδρα Οκάμπη που αντικαθιστά τον κύριο Βοσίσκη και για την Κούε η Σοφή Παλατιέ που αντικαθιστά τον ε, Ερνάντο Βαρένα. Αυτά λοιπόν είναι τα αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ψηφίσουν για λογαριασμό των τακτικών μελών. Επίσης να διευκρινίσω ότι Όλε οι πολιτικέ ομάδε θα πρέπει να ενημερώσουν τον προσωρινό πρόεδρο, εμένα δηλαδή, ε, σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε αλλαγή προτού ξεκινήσει η ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν τώρα στην διαδικασία ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο, ε, σε ό,τι αφορά την απαρτία. Διαπιστώνω ότι έχουμε περισσότερα από 17 μέλη και κατά συνέπεια έχουμε πλέον απαρτία και τώρα ζητώ να οριστούν οι υποψήφοι για την θέση του Πρόεδρου. Ε, παρακαλώ κύριο Ευχαριστώ, Κλοντ. Εκ μέρους των σοσιαλιστών ε, προτείνουμε τον Χωάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ ως ε, πρόεδρο, ο οποίος έχει ήδη θετεύσει το παρελθόν ως πρόεδρος της Επιτροπής. Καλώς λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, έχουμε ως υποψήφιο, έχουμε τον Χωάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ. Υπάρχει κάποια άλλη υποψηφιότητα. Έχουμε λοιπόν ένα υποψήφιο, Κουάν Φερνάντο Λόμπε Αγγιλάρ. Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η σημερινή μας συνάντηση είναι αφιερωμένη στη σύνθεση του προεδρίου της Επιτροπής μας. Η δικιά μου ομάδα δεν υποβάλλει υποψηφιότητα. Επιθυμία μου όμως είναι να μην ονομάζεται ε, πολιτικών ελευθεριών η Επιτροπή μας, αλλά μετανάστευσης, γιατί είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο απασχολεί τους λαούς μας, τα έθνη μας και είναι πολύ σημαντικό να ορίζονται τα θέματα τα οποία διακυδεύονται στην Επιτροπή αυτή και στον τίτλο. Ευχαριστώ πολύ. Μία υποψηφιότητα λοιπόν έχουμε. Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Όχι. Ωραία, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε. Ή μυστική ψηφοφορία Α, συγγνώμη. Προηγουμένως πρέπει να ρωτήσω, λέει ο Πρόεδρος. Έτσι είμαστε ε, ελευθεριών του πολίτη, η Επιτροπή. Οπότε πρέπει να ρωτήσω τον υποψήφιο. Δέχεται, δέχεται, Χουάν Δέχεσαι να αναλάβεις, να σου αφήσω την Προεδρία. Ναι, ναι, δέχομαι. Είμαστε μια ιδιαίτερη επιτροπή, οπότε πρέπει να σε ρωτήσω. Και να σου πω ότι χαίρομαι. Από τα πιο έμπειρα μέλη που μπορούν να αναλάβουν επίσημα την Προεδρία αυτή της Επιτροπής, έχοντας πείρα και στο Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας σου. Χαίρομαι λοιπόν διαβοή εγκρίνουμε τον Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ ως πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Um, Πολύ χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να δηλώσω τον Χουάν Φερνάντο Λόπες Άγγιλαρ εκλεγμένο πρόεδρο διαβοής της Επιτροπής μας. Χουάν, παρακαλώ, έλα να αναλάβεις τα καθήκοντά σου εδώ στη θέση του Πρόεδρου. Good afternoon everybody and first thing... Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από βάθος καρδίας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή για μένα που αναλαμβάνω και πάλι την Προεδρία της Επιτροπής αυτής. Ήμουνα παλιά το 2009 και τότε ήδη κατάλαβα ότι ήταν η πιο δραστήρια Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τεράστιο φόρτο εργασίας. Έχουμε πάρα πολλά επίκαιρα θέματα που συζητάμε στην Επιτροπή μας και κυρίως καλούμεθα να νομοθετήσουμε. Πολύ σωστά τα είπε ο Κλοντ. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος να βρίσκεται κανείς η Επιτροπή αυτή. Και για αυτούς που είναι από παλιά μέλη εδώ, εντάξει το ξέρουν, αλλά οι νέοι θα το καταλάβετε και από μόνοι σας πολύ σύντομα, ότι είναι μια εκπληκτική Επιτροπή αυτή. Γιατί χειρίζεται πολύ ζωτικά πολιτικά θέματα. Το επίπεδο το τεχνικό είναι επίσης ιδιαίτερα υψηλό σε αυτή την Επιτροπή και οι απαιτήσει είναι τεράστιες από κάθε άποψη. Γι' αυτό λέω ότι είναι τιμή μου ή ήταν τιμή μου όταν πρόεδρευα την πρώτη φορά. Ήταν ε, τιμή μου που με διαδέχτηκε ο Κλοντ Μωράης, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έμεινε πολύ στην ε, κεφαλή της Επιτροπής αυτής. Και ελπίζω να παραμείνει στην Επιτροπή μας για πολλά χρόνια ακόμα ο Κλοντ Μωράες. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας, Κλοντ. Και βέβαια και πάλι είναι μεγάλη μου τιμή που διαδέχομαι εγώ τον Κλοντ. Σας καλωσορίζω όλους στο έργο το οποίο θα αναλάβουμε. Είναι μια νέα αρχή και πάντα στην αρχή της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαστε γεμάτοι ελπίδες και φιλοδοξία. Να ξέρετε ότι είναι βούλησή μου να εξυπηρετήσω την Επιτροπή μας όσο γίνεται καλύτερα και στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, αλλά και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ξέρετε ότι θα φροντίσω να σας εκπροσωπώ όσο γίνεται καλύτερα και όσο μπορώ καλύτερα. Πάντα θα είμαι υπέρ των δικαιωμάτων της Επιτροπής αυτής επίσης στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Κάθε φορά που συζητάμε για τις δράσεις της δικής μας Επιτροπής η αφοσίωσή μας είναι τεράστια στο κράτος δικαίου, στα δικαιώματα των πολιτών, στην ηθαγένεια, τη μετανάστευση, την πολιτική ασύλου, εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασφάλεια, δικαστική συνεργασία, τόσο σε αστικά όσο και σε ποινικά ζητήματα, συνεργασία ε, αστυνομικών δυνάμεων για την καταπολέμηση ε, του διασυνοριακού εγκλήματος. Όντως λοιπόν είναι εκπληκτικό μέρος η Επιτροπή αυτή για να βρίσκεται κανείς και θα το δείτε ότι με ιδιαίτερη χαρά θα προεδρεύσω και θα σας εξυπηρετήσω εδώ από τη θέση αυτού και θα υπηρετήσω τις αρμοδιότητές μας. Λοιπόν, τώρα, για αυτήν την συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής μας. Ξέρετε ότι βάσει του άρθρου του κανονισμού 213 θα ψηφίσουμε για τέσσερις αντιπρόεδρους. Θα ψηφίσουμε όλους με την ίδια διαδικασία. Πρώτα λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε υποψηφίους για τις τέσσερις αυτές ε, θέσεις. Πρώτη αντιπροεδρία. Υπάρχει απαρτία, το έχουμε ελέγξει αυτό, να ξέρετε. τα τακτικά μέλη, οι αναπληρωτές που αντικαθιστούν τακτικά μέλη είναι επίσης εδώ και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου ή της πρώτης αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Οι υποψηφιότητες πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω ονόματα υποψηφίων. Παρακαλώ, είδα ένα χέρι εκεί. Παρακαλώ. Η κυρία Χετβέλτ. Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά, εκ μέρου ε, τη ομάδα Renew, προτείνω την κυρία Μάιτε Μπακαθαουρτουντούα. Ευχαριστώ για την πρότασή σας, κυρία Χιτφέλτ. Πρέπει να μου πει υποψήφια, πρώτον ότι συμφωνεί με την υποψιότητα και δεύτερον ότι έχει καλύψει τις προϋποθέσεις που είναι η δήλωση δεοντολογίας και οικονομικών συμφερόντων. Ναι, συμφωνώ. Δέχεστε λοιπόν τον ορισμό. Ωραία. Τώρα ρωτάω, υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες για αυτή τη θέση. Υπάρχει κανένα χέρι που σηκώνεται κάπου. Όχι, από ό,τι βλέπω. Συνεπώς, προτείνω διαβοής να εγκρίνουμε τον ορισμό αυτόν. So, I kindly request... Παρακαλώ την κυρία Ορτούντο να έρθει εδώ στο βήμα και να καθίσει. Παγκάσο Ορτούντο. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Το ίδιο ισχύει για θέση του Δευτέρου Αντιπρόεδρου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Τα μέλη είναι εδώ και περιμένω κάποιον να προτείνει υποψήφιο. Βλέπω να σηκώνεται κάποιο χέρι, έχετε το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε εν ονόματι της ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία θέλω να θέσω την υποψηφιότητα του Ζαν Μπολγκαρό. Θα ήθελα να σας πω το βιογραφικό του, διότι να δείξω που έχει επαγγελματισμό και εμπειρία. Και αυτά είναι χέγγια για την μελλοντική του θητή Ο Ζαν Πολγκορό είναι δικαστής και μέλος Εθνοσυνελεύσεως της Γαλλίας για 10 χρόνια και ασχολήθηκε με διάφορα θέματα παρόμοια με αυτά με τα οποία αυτή η Επιτροπή. Εκτέλεσε διάφορα καθήκοντα στο δικαστικό τμήμα στη Γαλλία. Δικαστή εισαγγελέα, πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αντιπρόεδρο τη Εθνική Σχολή ε, Δικαστών, αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου των ε, Παρισίων και σύμβουλο στον πρόεδρο τη ε, Γερουσίας έχει εμπειρία επαγγελματική, κοινοβουλευτική και μπορεί να εκτελέσει με έξοχο τρόπο αυτά τα καθήκοντα. Ε, και τον προτείνουμε για την εκλογή του. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ταρντίνο, για την πρότασή σας. Άλλη υποψηφιότητα έχουμε. Βλέπω κάποιο χέρι. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Να προτείνω για θέση δευτέρου αντιπροέδρου τον Πιέτρο Μπάρτολο, τον Ιταλό συνάδελφό μα. νέο μέλος στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο, αλλά έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, εργαζόμενος επιτόπου στη Λαμπεντούζα, στην Ιταλία, όχι μόνο για θέματα μεταναστών, αλλά σε διάφορους τομείς. Αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι ένα από τα μέλη του Κοινοβουλίου με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων που τον εξέλεξαν. Θα ήταν πολύ καλό να τον έχουμε στη θέση του Αντιπροέδρου και να εκπροσωπεί την ομάδα μας σε κάποιους από τους σημαντικότερους τομείς που πρέπει να επεξεργαστούμε σε αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελ. Έχουμε δύο υποψηφίους. Άλλος υπάρχει, άλλη υποψηφιότητα, άλλη πρόταση. Θα κάνουμε το εξής λοιπόν. Θα ρωτήσω και τους δύο υποψηφίους αν δέχονται την υποψηφιότητά τους, αν συνενούν και αν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για να γίνουν αντιπρόεδροι. Ο κ. Ζαν Πολ Ζαγότ, δεχόσαστε την υποψηφιότητα, τη δέχομαι κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Έχετε συμπληρώσει τα, αυτή τη δήλωση για οικονομικά συμφέροντα και την δήλωση για τα διοντολογικά θέματα. Όλα, όλα. Σας ευχαριστώ. Έχουμε δεύτερο υποψήφιο. Ε, συνάδελφε Μπάρτολο, δέχεστε την υποψηφιότητα. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Μπάρτολο. Συμπληρώσατε και τη δήλωση για οικονομικά συμφέροντα και για την ε, καλή συμπεριφορά, τα δεντολογικά θέματα. Έχουμε δύο υποψηφίους που έχουν αποδεχθεί την υποψηφιότητά τους. Άρα, τώρα πρέπει να ψηφίσουμε μέσω μυστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Έχουμε τις κάρτες, οπότε θα αρχίσουμε σε λίγο την ψηφοφορία. Αν έχετε όλοι τις κάρτες σας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε γιατί είναι αποφασιστική σημασία. Να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε μια κάρτα και έχουμε και το μηχανηματάκι με τρία κουμπιά. δεν θα είναι μυστική ψηφοφορία. Αλλά πρέπει να πατήσετε ένα κουμπί για κάθε υποψήφιο της προτιμήσεώς σας. Με αλφαβητική σειρά, το πρώτο κουμπί είναι για τον κύριο Μπάρτολο. Το δεύτερο κουμπί για τον κύριο Ραγό. Το κόκκινο κουμπί, με άλλα λόγια, είναι ψήφος υπέρ του κυρίου Μπάρτολο. Και το κόκκινο κουμπί. Αλφαβητική σειρά. Δεν σημαίνει το κόκκινο είναι αρνητικό. Είναι ψήφο υπέρ του κυρίου Ραγό. Είναι θέμα του να πατήσετε ένα κουμπί για κάθε υποψήφιο που θέλετε. Για να δούμε ποιο θα είναι ο νικητής. Μόνο αυτό το νόημα έχει. Η κυρία Έντφελτ κατανοώ. Κάθε κουμπί είναι για ένα υποψήφιο. Μπορεί να είμαστε σαφεί όσον αφορά τα χρώματα. Ποιο κουμπί αφορά ποιον υποψήφιο, παρακαλώ. Τα χρώματα να μα καθαρίσετε. Μου είπαν από τη γραμματεία. Είναι αμερόληπτη επιλογή και δίκαιη. Σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά. Το B είναι πριν από το G. Μπάρτολο είναι πρώτο. Άρα πράσινο. Πράσινο κουμπί για τον Μπάρτολο και το κόκκινο για τον κύριο Γκαγό. Μόνο λόγω αλφαβητική σειρά. Μόνο έτσι γίνεται η επιλογή. Δεν σημαίνει το πράσινο είναι ναι και το κόκκινο είναι όχι. Θα είναι μυστική ψηφοφορία. Πράσινο για τον κύριο Μπάρτολο, κόκκινο για τον κύριο Γκαγόν. Εάν το κόκκινο έχει περισσότερου ψήφου από το πράσινο, ο κύριο Γκαγό, Γαγό είναι αντιπρόεδρο. Αν αντιστρόφω, ο κύριο Μπάρτολο θα είναι ο αντιπρόεδρο. και τέλος της ιστορίας. Αυτό θα κάνουμε. Ξεκάθαρο. Πράσινο, μπάρτολο. Κόκκινο, γκαγό. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. ωραία. Αν είναι ξεκάθαρο, συμφωνούμε. Η κυρία Σίπελ, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πράσινο ή κόκκινο κουμπί δεν είναι ναι ή όχι. Έχετε μόνο ένα ναι ένα κουμπί για ναι. Στην περίπτωση του κ. Μπάρτολο είναι πράσινο και στην άλλη περίπτωση είναι κόκκινο. Αν δεν θέλετε να ψηφίσετε έναν από του υποψηφίου, απλώ κάνετε τίποτα. Δεν πατάτε κανένα κουμπί. Σωστά. Αν δεν θέλετε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή, μπορείτε και να πόσχετε. Λευκό κουμπί με άλλα λόγια. Το λευκό κουμπί σημαίνει αποχή. Αλλά Πιστέψτε με τώρα που σας το λέω. Είναι μυστική ψηφοφορία. Δεν θα υπάρχει στη διάθεση σας κόκκινο ή πράσινο φως που θα ανάβει. Πάντα γαλάζιο φως θα ανάβει. Θα παραμείνει μυστική ψήφο σας. Αν στην οθόνη τα κόκκινα είναι περισσότερα από τα πράσινα, αυτό σημαίνει ότι ο κ. Γκαγό θα είναι αντιπρόεδρος. Αντίστροφα, αν πράσινε ψήφοι είναι οι περισσότερε από τι κόκκινε, ο κύριο Μπάρτολο. Αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν τον κύριο Μπάρτολο, πατήστε πράσινο. Εκείνοι που θέλετε να ψηφίσετε τον κύριο Γκαγό, πατήστε κόκκινο. Και εσεί θέλετε να πόσχετε, που έχετε δικαίωμα, πατήστε το λευκό κουμπί. Έτσι. Ωραία. Αν είναι ξεκάθαρο, α ξεκινήσουμε λοιπόν. Τώρα ξεκινάει η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ο κύριος Μπάρτολο. Κύριε Μπάρτολο, έχετε εκλεγεί αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Σας καλούμε να έρθετε εδώ, στο βήμα, για να συμμετάσχετε στο Προεδρείο. Ευχαριστώ όλους σας που ψηφίσατε. Ευχαριστούμε και τους υποψηφίους. Σαφές το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Καλούμε τον κύριο Μπάρτολο να έρθει εδώ. Πάμε τώρα για τη θέση τρίτου αντιπροέδρου, ακριβώς η διαδικασία. Περιμένουμε υποψηφιότητα. Η ε, κυρία Ματσόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, συγχαρητήρια από όλου μα. Προσβλέπουμε συνεργασία μαζί σα στη θητεία αυτή. Θέλουμε να, να προτείνουμε τον κύριο Μπάρασιτ για τη θέση τρίτου Προέδρου. Mr. Σιτβέγγι. Itvegi. Είσαστε, είσαστε εδώ. Δέχεστε την υποψηφιότητά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δέχομαι έχετε συμπληρώσει τα δέοντα, τις δηλώσεις κλπ. Συμπληρώσατε τα πάντα. Ωραία. Άλλη υποψηφιότητα. Βλέπουμε και, άλλη, και άλλο χέρι να σηκώνεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και από μένα προς εσάς και τους αντιπροέδρους που εξελέγησαν. Νταμιάν Καράν, τον υπέροχο συνάδελφο, την υπέροχη συνάδελφο προτείνουμε. τον κύριο Νταμιέν Καρεμέ. Προτείνουμε. Δέχεστε, κύριε Καρεμέ. Δέχομαι. Και έχω κάνει όλα τα τυπικά που έπρεπε να συμπληρώσω. Λέτε ναι και έχετε συμπληρώσει τη δήλωση, έχετε ολοκληρώσει τις τυπικές διαδικασίες. Έχουμε δύο υποψηφιότητε. Άλλος, ορίστε, κύριε Ματσόλα, παράλλα Βλέποντα την κατάσταση, πρέπει να διαβουλευτώ με του άλλου συντονιστέ και του συναδέλφου και ζητώ να διακοπεί υπό τι περιστάσει η συνεδρίαση. Λογικό αυτό, σα πειράζει να το κάνουμε αυτό, να διακόψουμε. Ε, για πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεστε. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, γι' αυτό χρειάζομαι μερικά λεπτά. Πέντε λεπτά φτάνουν. Ωραία. Αν δεν σας πειράζει, εφόσον υπάρχει μία διέξοδος από ό,τι φαίνεται από αυτό τον ανταγωνισμό αν θέλετε ας διακόψουμε 5 λεπτά και σε 5 λεπτά θα συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες της Επιτροπής. Ευχαριστώ.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 Συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κατανοούμε την κατάσταση. Please take your seats. Παρακαλώ καθίστε. I may call your attention, Madame Madame Reike. Κυρία Ματσόλα, κυρία Ράικε, κυρία Σίπελ, σας παρακαλώ. Κυρία Εντφέλτ. Madame Ernst. I understand that there are the coordinators involved. οι συντονιστές ας βοηθήσουν. Ας περιμένουμε λίγο να έρθουν οι συντονιστές, να συνεννοηθούν. Καθίστε, νομίζω ότι υπάρχει διέξοδος. Η κυρία Ματσόλα τι έχει να πει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας. Προτείνω και ελπίζω να υποστηρίξουν συνάδελφοί μου σε αυτό, να διακόψουμε την εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου σε αυτή την επιτροπή. Το ίδιο έγινε και σε άλλε επιτροπέ για παρόμοιου λόγου. Και αν επιτρέπετε όμω να πάμε στην εκλογή του τέταρτου αντιπροέδρου, ούτω ώστε το ΕΛΚ να έχει έναν εκπρόσωπο στο παρόν Προεδρείο, ενώ η θέση του τρίτου αντιπροέδρου εξετάζεται. Κατανοώ, κατανοώ. Και βλέπω ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία όσον αφορά αυτό το αίτημα. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο, δίκαιο αίτημα διότι θεωρούμε ότι το ΕΛΚ είχε την επιλογή υποβολής υποψηφιότητας, θέλουν να το ξανασκεφτούν, αν προχωρήσουμε για τη θέση του τετάρτου αντιπροέδρου, ξεκαθαρίζει η κατάσταση με δίκαιο τρόπο και θα περιμένουμε από το ΕΛΚ μια κάποια αντίδραση. Σηκώνεται κάποιο χέρι. Η κυρία Σίπελ, θέλετε να πείτε κάτι. Συμφωνώ με την πρόταση και να κάνουμε την ψηφοφορία του τέταρτου αντιπρόεδρου και ελπίζω μετά οι ομάδες να βρουν μια λύση για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Κι άλλο χέρι. Έχετε το λόγο. Εγώ είμαι κατά να γίνει ψηφοφορία τώρα του τετάρτου αντιπρόεδρου, γιατί από την εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου θα εξαρτηθεί η εκλογή του τέταρτου αντιπροέδρου. Δηλαδή μετά από την τρίτη θα, από τρίτη εξαρτηθεί η τέταρτη ε, ε, ψηφοφόρια. Οπότε εγώ θα ε, πρότεινα να συνεχίσουμε με την εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου ή να αναβάλουμε συνολικά τις υπόλοιπες ψηφοφορίες. Ε, εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με αυτή τη λύση. Δηλαδή και εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε τώρα να προβούμε στην εκλογή του τετάρτου αντιπροέδρου και από εκεί και μετά να να στείλουμε για αργότερα την εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Να ε, την αναβάλουμε. Δηλαδή νομίζω πως ε, είναι μια λύση η οποία είναι βιώσιμη. Κυρία Και κυρία Ίντβελτ κάτι θέλει να πει. Ναι. Στηρίζουμε το αίτημα για αναβολή. Δεν μας αρέσει πολύ, είναι ατυχής η κατάσταση. Η αναβολή ζητήθηκε από το ΕΛΚ για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Ελπίζω το ΕΛΚ επίση να υπομειστεί τις ευθύνε του και να εξασφαλίσει ότι όταν ψηφίζουμε σε 10 μέρες ότι θα έχει βρεθεί μια λύση και δεν θα ξαναβρεθούμε σε μια παρόμοια κατάσταση. Άλλος, έχει το λόγο. Εμείς από τους Πρασίνους δεχόμαστε την πρόταση αναβολής της ψηφοφορίας και όπως είπε η κυρία Ιντφέλτ ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί μια λύση στο χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη ψηφοφορία. Και υποστηρίζουμε και την άλλη πρόταση να ψηφίσουμε τώρα για τη θέση του τετάρτου αντιπρόεδρου. Καλώς, πλευρά Προέδρου, σας ευχαριστώ για την κατανόησή σα. είναι απροσδόκητη αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και προτάθηκε μια διέξοδο, ενδεχόμενη διέξοδο. Πρώτα από το συντονιστή, ε, την κυρία Ματσόρα, τη συντονίστρια του ΕΛΚ που έχει τον πρώτο λόγο. Και σαν προέδρο βλέπω ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια πλειοψηφία που υποστηρίζει αυτή την πρόταση τη κυρία Ματσόλα. Δηλαδή, οι συντονιστέ των μεγαλύτερων ομάδων τη ε, Επιτροπής υποστηρίζουν αυτή την πρόταση. Η θέση τρίτου αντιπροέδρου, η ψηφοφορία, η θέση τρίτου αντιπροέδρου να αναβληθεί και να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία για θέση τετάρτου αντιπροέδρου. Και αυτό θα κάνουμε τώρα. Θέση τετάρτου αντιπροέδρου. Να δούμε ε, ποιες υποψηφιότητες έχουμε. Ε, κυρία Ματσόλα, ευχαριστώ. Η ομάδα του ΕΛΚ. Τον κύριο Έμιλ Ράντεφ προτείνει για αυτή τη θέση. Βετεράνος και αυτός Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Δέχεστε. Δέχεστε. Έχετε συμπληρώσει τα έντυπα που πρέπει, τις τυπικές διαδικασίες, τα πετούμενα έγγραφα. Ναι. Καλώς, άλλη υποψηφιότητα. Υπάρχει. Δεν βλέπω. Εν τη αυτή περιπτώσει μπορούμε διαβοής να σας ανακηρύξουμε μέλος του Προεδρείου. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Ράντεφ.

Άλλο ένα λεπτάκι για να τελειώσουμε αυτή τη συνεδρίαση στάσεως σε σώμα τη Επιτροπή μα Ευχαριστώ όλου εκ βάθου καρδίας. Προσωπικώ σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και μιλώ και εκ μέρου των άλλων μελών του Προεδρείου. Αύριο, ανακοινώσει του Προέδρου, αύριο θα έχουμε πρώτη συνεδρίαση συντονιστών. στις 10. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη συνεδρίαση συντονιστών. Και συνεδρία συντονιστών θα υπάρχει περιθώριο για επίλυση της εκκρεμότητας της θέσης του τρίτου αντιπροέδρου. Θα έχουμε περισσότερα περιθώρια λιγμών για το ΕΛΚ. Και η συντονίστρια κυρία Ματσόλα θα έχει σε λιγμών για να βρει επικοδομητική λύση για την ώρα. Θα γιορτάσουμε την πρώτη συνεδρίαση, την ε, τακτική συνεδρίαση. Μάλλον θα αρχίσουμε την πρώτη τακτική συνεδρίαση την εβδομάδα στις 20, μετά το Στρασβούργο, 24-25 ε, Ιουλίου. Καλείστε να συμμετάσχετε στην πρώτη τακτική συνεδρίαση.